Τα συνοπτικά πρακτικά τη χθεσινή συνεδρίαση και τα κείμενα που εγκρίθηκαν κατά συνεδρίαση αυτή έχουν διανεμηθεί. Υπάρχουν παρατηρήσει. Δεν βλέπω κανέναν. Τα συνοπτικά